η συζήτηση. You started the day with me, you ended with me. Κλήγη συνεδρίαση. Ξεκίνησε με μένα, λίγη με μένα, λέω